πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση για τα χρηματοδοτικά μέσα και μάλιστα έχουμε πολλές εκθέσεις. Πρώτα απ' όλα η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Γκέρενς για το μηχανισμό, μηχανισμό χρηματοδότηση αναπτυξιακή συνεργασία. Μετά, σύσταση για δεύτερη ανάγνωση των κυρίων Λόχμπιλε και Γκάλ. Χρηματοδοτικό μέσο για την παραγωγή τη δημοκρατία και των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατόπιν σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Μίτσελ, μηχανισμός χρηματοδότησης αναπτυξιακής συνεργασίας και σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Σόλτς, θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Πρώτα απ' όλα θα λάβουν το λόγο όλοι οι εισηγητές και πρώτα απ' όλα ο κύριος Γκέρνς για 4 λεπτά. Παρακαλώ. Το σχέδιο κανονισμού που συστήνει ένα μηχανισμό συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα για τις χώρες ΑΚΕ εξετάζεται σε δεύτερη ανάγνωση σήμερα. Σας πενθυμίζω ότι στην πρώτη ανάγνωση ταχθήκαμε υπέρ των μέτρων που θα βοηθήσουν τις χώρες που εξάγουν μπανάνα